προτάσεις να σας κάνω. Τα χαρτιά μου είναι στα τσεχικά και θα τα διαβάσω τσεχικά. Θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία Ζανίν Χένις Πλάσχαρτ και ο κύριος Πακέ μας διαβίβασαν γραπτός ότι ε, ε, παρετούνται από το αξιώμα του Ευρωβουλευτού ε, διότι εξελέγησαν στη Βουλή των κάτω χωρών. Και